θέσεως Μαρίνιο Επίντο για το ΔΕΚ της Ευρωπαϊκής Ενώσεως αριθμός των δικαστών θα δώσω το λόγο του, τον εισηγητή Παρακαλώ σεβαστείτε το χρόνο αγόρευσης Σε ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2011 ξεκίνησε μια νομοθετική πρωτοβουλία για την τροποποίηση του καθεστώτος ώστε να μπορέσουν να εκλεγούν επιπλέον 12 δικαστές στο Γενικό Δικαστήριο. Τον Απρίλιο του 2014 έτυχε σε πρώτη ανάγνωση έγκριση του Ευρωκοινοβουλίου. Ωστόσο το Συμβούλιο δεν διόρισε κανέναν από αυτούς τους 12 ε, δικαστές ε, και δεν κατάφεραν να συνεννοηθούν στην επιλογή των δικαστών αυτών τα κράτη-μέλη κάθε κράτος ήθελε να διορίσει το δικό του δικαστή και ο αριθμός των δικαστών που θα διοριζόντουσαν 12 δεν ανταποκρινόταν στον αριθμό των κρατών που θα επέλεγαν 28. Και έτσι λοιπόν το 2014 ζήτησε το δικαστήριο επιπλέον 28 ε, δικαστές. Δηλαδή πάνω από το, ε, ζήτησε τον διπλασιασμό του αριθμού των δικαστών του Γενικού Δικαστηρίου. Τον Απρίλιο, το, το, το, το προηγούμενο έτος επαρκούσαν 12 δικαστές μετά στη συνέχεια απαιτούνται ξαφνικά 28 δικαστές ε, μετά από ε, δράση του δικαστηρίου. Είναι προφανές ότι δεν πρόκειται να λυθεί έτσι κανένα πρόβλημα του δικαστηρίου. Είναι η αναζήτηση λύσης του Συμβουλίου για την επιλογή του αριθμού των δικαστών για να ανταποκρίνεται ο αριθμός αυτός στον αριθμό των μελών του Συμβουλίου. Δεν πρόκειται εδώ λοιπόν απλά για μια αλλαγή σε μια νέα πρόταση. Πρόκειται για μια απόλυτα νέα πρόταση. Όχι μόνο 12 βουλευτές αλλά επιπλέον 28 βουλευτές που απαιτούνται και ενός εξειδικευμένου δικαστηρίου που προβλεπόταν και από, το, ε, από τη συνθήκη της Τώρα η νέα νομοθετική αυτή πρόταση σύμφωνα με αυτήν η Επιτροπή θα έπρεπε υποχρεωτικά να τοποθετηθεί επί του περιεχομένου της πράγμα το οποίο δεν, δεν συνέβη. Ε, τοποθετήθηκε για την επιλογή επιπλέον 12 δικαστών και όχι για τους 28 βουλευτές και δεν γνωμοδότησε για αυτή την τοποθέτηση του ε, δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι συνθήκες ζητούν εξειδικευμένα δικαστήρια και όχι την κατάργησή τους. Αυτό θα σήμαινε την ε, εγκατάλειψη του συστήματος των εξειδικευμένων δικαστηρίων που προβλέπονται από τη συνθήκη της Λισαβόνας. Ενώ γνωρίζουμε ότι η εξειδικευμένη δικαιοσύνη είναι δικαιοσύνη αναβαθμισμένης ποιότητας και δυνατοτήτων. Γι' αυτό θα έπρεπε νέα δικαστήρια εξειδικευμένα να δημιουργηθούν, ιδιαίτερα για τα διπλώματα ευρεσιτεχνία και τις μάρκες, ε, για να μπορούν έτσι να είναι αποτελεσματικά. Μια μεταρρύθμιση αυτή τη φύση θα έπρεπε να προηγείται από μια μελέτη επιπτώσεων που οι συνομοθέτες Συμβούλιο και Κοινοβούλιο θα γνωρίζουν τα σχετικά με τις επιπτώσεις, το κόστος και όλες τις ε, συνέπειες. Πράγμα το οποίο δεν έγινε. Και για την ε, πρόταση του Συμβουλίου προτείνω στην έκθεσή μου την αποκατάσταση αυτού που ενέκρινε σε πρώτη ανάγνωση του, το Κοινοβούλιο τον Απρίλιο του 2014 να ξαφνικά να περάσουμε από τους 12 δικαστές στους 28 δεν θα το κατανοούσαν ποτέ οι πολίτες μας. Μια και θα σήμαινε τεράστια αύξηση των δαπανών, πάνω από 100 εκατομμύρια ευρώ. Απλά και μόνο επειδή δεν μπόρεσε το Συμβούλιο να επιλέξει τους αναγκαίους δικαστές. Σε μια περίοδο όπου πλήττουν αυστηρά μέτρα λιτότητα στις χώρες μας και προτείνεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση περικοπή των δημόσιων δαπανών να αυξήσουμε έτσι τις διαθροτικές δαπάνες της Ευρωπαϊκής θα ήταν πολύ αρνητικό παράδειγμα για το σύνολο της Ευρώπης. Όμως το Συμβούλιο δεν ακολούθησε αυτή τη σκέψη και αυτά τα επιχειρήματα. Διατηρεί αυτή τη λογική τη δική του και θέλει να διπλασιαστεί ο αριθμός ε, των ε, δικαστών. Η δική μου ε, έκθεση ζητεί απόλυτη κατά το ίμιση σύνθεση ανδρών και γυναικών των μελών του δικαστηρίου. Αλλά και πάλι εδώ δεν ακολουθείτε αυτή η πρόταση από το δικαστήριο. Μία δήλωση υποβάλλεται χωρίς καμία νομική δεσμευτική υποχρέωση. Θα πρέπει λοιπόν στην Ευρωπαϊκή Ένωση να, θεωρήσουμε ότι δεν περνάει η ισότητα των φύλων μέσα από ε, δηλώσεις. Πρέπει λοιπόν ε, μέσω του συνταγματικού δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης να θεωρήσουμε ότι δεν επιτρέπεται η υλοποίηση ενός ε, θεμελιώδους συνταγματικού δικαιώματος. Και για αυτόν τον λόγο ακόμα Ακόμα απαιτώ την απόρριψη της θέσης του Συμβουλίου και την επιστροφή στο αποτέλεσμα της πρώτης ανάγνωσης από το, Ευρωκοι... από το Ευρωκοινοβούλιο. Το λόγο τον έχει η κυρία Κρετσού. Από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κύριε Σιγητά, αγαπητοί συνάδελφοι, υποστηρίζει τη συμβιβασμό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τη συμβιβασμό μεταξύ Συμβουλίου και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αυτό ο συμβιβασμό είναι αποτέλεσμα μακρών διαπραγματεύσεων και πετυχαίνει ισορροπημένη λύση. Η λύση μας επιτρέπει να προχωρήσουμε επί ενός θέματος που είχε αποτελεματωθεί επί μακρόν. Θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας επίσης ότι ο συμβιβασμός άμεσα εδράζεται επί ιδεών που έχουν υποβληθεί από το ΔΕΚ το ίδιο. Θα πρέπει να ολοκληρωθεί μεταρρύθμιση. Είναι πολύ σημαντικό αυτό κατά την άποψή μας η κατάσταση εντό του Γενικού Δικαστηρίου παραμένει πηγή ανησυχιών. Αυτή η μεταρρύθμιση θα επιτρέψει στο δικαστήριο να μειώσει τι καθυστερήσει όσον αφορά την εκδίκαση των υποθέσεων και θα επιταχύνει τις διαργασίες του. Αποτελεσματική δικαστική αναθεώρηση είναι θεμελιώδες δικαίωμα, το οποίο το εγγυάται η χάρτα. Όμω, η αναθεώρηση δικαστική είναι αποτελεσματική αν είναι και έγκαιρη. Το χρωστούμε λοιπόν στου πολίτε αυτό και στους οικονομικούς φορείς. Πρέπει να ενισχύσουμε τις δυνατότητες που έχει το δικαστήριο, να μπορεί να εκδικάζει γρήγορα τις υποθέσεις. Ταχεία διευθέτηση των διαφορών, των νομικών, είναι υποφελής για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και για την Ένωση στο σύνολό της. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επίσης καλωσορίζει τη λύση που εξευρέθη, δηλαδή να προωθηθεί ισορροπία των φύλων εντός του δικαστηρίου. Είναι κοινό στόχος, αντικειμενικός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Να υποστηρίξω λοιπόν την πλήρη υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον Πτευθέντα Συμβιβασμό και αν εγκριθεί τελικά το κείμενο θα τοποθετηθούμε θετικά επί των τροπολογιών, αν αυτές εγκριθούν και από τις συζητήσεις που θα διεξαχθούν. Ξεκινάμε λοιπόν τον γύρο των ομάδων. Ο κύριος Τσέφκα έχει το λόγο επί δύο λεπτά εν ονόματι του ΕΛΚ. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, κυρία Επίτροπε, μια λειτουργούσα δικαιοσύνη είναι ένας από τους πιο σημαντικούς πυλώνες ενός δημοκρατικού κράτους και η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια οικογένεια δημοκρατικών κρατών. Γι' αυτό πρέπει να λειτουργεί εύθετα και σωστά η ευρωπαϊκή δικαιοσύνη. Και αυτό είναι κάτι που υποστηρίζουμε όλοι μα. Για αυτού του λόγου θέλω εξ ονόματο του ΕΛΚ με μεγάλη ικανοποίηση να δηλώσω ότι μετά από μακροχρόνιε διαπραγματεύσει τώρα καταλήξαμε σε, καταλήγουμε σε έναν συμβιβασμό. Και έχουμε διαπραγμάτευση συμβιβαστικών προτάσεων μεταξύ του Ευρωκοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Αυτός ο συμβιβασμός θεμελιώνεται στην αναγνώριση της αναγκαιότητας της αύξησης του αριθμού των δικαστών στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Γνωρίζουμε ότι πρέπει να αυξηθεί ο αριθμός των δικαστών στο Ευρωδικαστήριο για να λειτουργεί καλύτερα και να είναι πιο αποτελεσματικό. Και δεν πρέπει να είναι ιδιαίτερα ε, χρονοβόρες ε, οι εξεταστικέ διαδικασίε από το Ευρωδικαστήριο Δικαστήριο. Κατάφερε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εισαγάγει δύο στοιχεία. Έχουμε τώρα τη δυνατότητα μετά την ολοκλήρωση των μεταρρυθμίσεων να επανεξετάσουμε και να δούμε ποια είναι η κατάσταση πραγμάτων και ποιο αποτέλεσμα επετέφθη στην λειτουργία συνολικά του Ευρωδικαστηρίου ανάλογα με αυτά τα οποία επιθυμούσαμε και είχαμε ως φιλοδοξίες. Δεύτερον, υπάρχει ένα ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου από κοινού με το Συμβούλιο όπου γίνεται αναφορά στην ανάγκη, στην αναγκαιότητα να υπάρχει εξίσωση των ε, φύλων, του αριθμού των δικαστών όσον αφορά τα δύο φύλλα. Και θα πρέπει αυτή η αναλογία να ε, θεσπίζεται και να ισχύει σε όλα τα θεσμικά όργανα και όχι μόνο σε ένα. Είναι μακρά η πορεία και εξ ονόματος του ΕΛΚΑ υποστηρίζω εγώ και υποστηρίζουμε εμείς αυτό το συμβιβασμό και το Συμβούλιο. Ευχαριστώ. Έχουμε σοσιαλιστών η κυρία Ντελβό. Έχει το λόγο για ένα λεπτό. Merci. Ε, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η δικαιοσύνη είναι μια θεμελιώδης αρχή, ένα δικαίωμα και μια υποχρέωση καθήκων μέσα σε μια δημοκρατία και η δικαιοσύνη της Ένωσης ε, βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε δυσκολία. Ως εκπρόσωπος των, πολιτών, εκπρόσωποι μάλλον των πολιτών, πρέπει να την υπερασπιστούμε δίνοντάς της τα μέσα που χρειάζεται για να μπορεί να ελοποιεί το έργο της. Ε, υπάρχει έλλειψη, αυτό είναι ένα φίβολο. Τα οι υποθεσει υποθέσεις ε, αυξάνονται από έτος σε έτος και οι προσφυγές για μη σεβασμό της προθεσμίας ε, έχουν επίσης πολλαπλασιαστεί και το κόστος τους ανέρχεται στα 27 εκατομμύρια, δηλαδή μέγα κόστος δεν θα πρέπει να αφήσουμε να περάσει αυτή η ευκαιρία να επιτύχουμε ένα στόχο για την ισότητα των φίλων που πολλές φορές έχει αναφερθεί στις ε, συμβολικές δηλώσεις. Γι' αυτό και καλό όλους τους δημοκράτες να υπερψηφίσουν αυτή την πρόταση για μεγαλύτερη ισότητα και δικαιοσύνη μέσα στο ΔΕΚ. Ε, δέχεστε μπλε κάρτα από τον κύριο Σιλ. Δεν μας έχει πει. Ο κύριος Πόσπης χωρίς μικρόφωνο. Μάλιστα. Και εδώ πρέπει να αναφερθώ στο ότι υπάρχουν προβλήματα με όλο και περισσότερες περιπτώσεις και θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με την πρόσληψη νέων ε, δικαστών. Έτσι θα πρέπει να το δούμε. Euh, ναι, καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι το να έχουμε πολλούς ε, ε, καταγγέλλοντες ανα, αναδικαστεί, αυτό οδηγεί σε, σε, μη, σε μη δυνατότητα διεκπαιρέωση των υποθέσεων. Θα πρέπει να τους δώσουμε περισσότερη βοήθεια. Κυρία Πρόεδρε, κύριος Καρύμ, 20 χρόνια ε, υπηρετώ τους ε, ψηφοφόρους. Εδώ υπάρχει μεγάλη κολλησιεργία. Το υπήρξα μάρτυρας αυτού μέχρι τώρα. Δεν τα λέω έτσι ελαφρά την καρδία. Έχω εμπλακεί στην ε, νομική επιτροπή συνεργαζόμενος με συναδέλφους μαζί με τον εισηγητή προσπαθώντας να βρούμε σωστή λύση για το παρουσιαστέν πρόβλημα. Όμως, για μία ακόμη φορά, μία πραγματική ευκαιρία για μεταρρύθμιση δεν οδηγήσε στη σωστή προσέγγιση. Παραδώσαμε αυτή την ευκαιρία, τη θυσιάσαμε στο βωμό της πολιτικής ε, προσέγγισης, να προχωρήσουμε γρήγορα προς μία λύση που δεν είναι λύση. Όλοι οι πολίτες Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτούν πραγματικές μεταρρυθμίσεις μεταρρυθμίσεις που αντικατοπτρίζουν οι υπηρεσίε που παρέχονται. Εμεί τη διαλέξαμε, για μία ακόμη φορά διαλέξαμε ένα συμβιβασμό. Μία λύση που προσθέτει στο άκθος των πολιτών και δεν κάνει τίποτα για την εξέβρεση λύσεως στα προβλήματα. Προβλήματα που μας παρουσιάστηκαν. Συνάδελφοι, θα δαπανίσουμε 20 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Παραπάνω ευρώ όταν δεν χρειαζόταν να προσθέσουμε ούτε σεντ στο βάρος για τους Ευρωπαίους φορολογουμένους. Συνάδελφοι, όλοι αποτυγχάνουμε στο στόχο μας. Γι' αυτό τι έκανα εγώ. Να προτείνω μια τροπολογία, ένα ψήφισμα που απορρίπτει τη θέση του Συμβουλίου. Και καλό τους συναδέλφους όπως μου είπαν κατηδίαν ότι γνωρίζουν και αναγνωρίζουν ότι τα επόμενα χρόνια θα λυπηθούμε και θα μετανιώσουμε για την απόφασή μας. Ζητώ λοιπόν να υποστηρίξουν τη δική μου πρόταση. Ο κύριος Καβαντά για 1,5 ε, λεπτό έχει το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Προέδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Το σχέδιο μεταρρύθμισης που εξετάζουμε τώρα και που διαπραγματευτήκαμε στον τριμερή διάλογο θα μας επιτρέψει να ασκήσουμε δημοσιονομικό έλεγχο αυξημένο όσον αφορά τις πραγματικές ανάγκες του ΔΕΚ και να παγιώσουμε μια απαραίτητη λειτουργία ύψης της δημοκρατίας. Δικαιοσύνη δηλαδή που τη ζητούν, τη διεκδικούν οι πολίτες. Μετά τη δημοσίευση της προτάσεως μεταρρυθμίσεως του 2012, ο αριθμός των υποθέσεων που εκδικά στο δικαστήριο αυξήθηκε κατά 43% το 2014. Πέντε ήδη προσφυγές κατετέθησαν για επέρβαση χρονικής διαρκείας, χωρίς να αποφασίσει η δικαιοσύνη. Και αυτό σε αποζημιώσεις κοστίζει 27 εκατομμύρια και σε τόκους. Τεράστια ζημία. Η μεταρρύθμιση λοιπόν είναι εξελικτική, διαθρωτική του δικαστηρίου που ζητείτε, την υποστηρίζω. Μας επιτρέπει αυτή η αλλαγή να έχουμε τρία στάδια. Και στο τέλος κάθε σταδίου υπάρχει μια αποτίμηση που πραγματοποιείται για να δούμε αν πρέπει να προχωρήσουμε πιο πέρα. Συνεπώ, δεν έχω κανένα φόβο όσον αφορά το επιχείρημα της οικονομικής ζημίας. Είναι δημαγωγικό επιχείρημα. Και να πω κάτι εν τέλει. Δεν, υποτιμούμε, δεν πρέπει να υποτιμούμε το δημοκρατικό λειτουργικό αυτό, διότι αν μοιάζει σαν κάτι, είναι σαν εκτελεστικός νομοθετικός κλάδος στα μάτια του ε, λαού και θα πρέπει να έχουμε και ένα δικαστικό κλάδο ο οποίο τελικά να λειτουργεί. Η κυρία Χάουταλα για τους πρασίνους. Για 1,5 λεπτό έχει το λόγο. Um, κυρία Πρόεδρε, βρισκόμαστε στη δεύτερη ανάγνωση αυτού του ζητήματος και από το 2011 το Συμβούλιο, σύμφωνα με τη δική μου εκτίμηση, ποτέ δεν πρόκειται και να ε, τροποποιήσει αυτή την ε, αίτημα για 28 νέους δικαστές. Αλλά για όσους αυτό το αμφισβητούν θέλω να υπογραμμίσω ότι αυτή η μεταρρύθμιση δεν αφορά μόνο τον αριθμό των δικαστών και την έρηδα που έχει ε, δημιουργηθεί γύρω από αυτό. Αυτό το θέμα αφορά την αποτελεσματικότητα του Ευρωπαϊκού Δικαστικού Συστήματος και είναι πολύ σημαντικό αυτό το σύστημα για την προστασία των πολιτών. Το δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι αυτό που προστατεύει το κράτος δικαίου, τη διαφάνεια και τα θεμελιώδη δικαιώματα. Η ποιότητα αυτού θα πρέπει λοιπόν να είναι η υψηλότερη μας προτεραιότητα. Στου τριμερείς διαλόγου στο Κοινοβούλιο έχει επίσης επιτύχει κάτι ιστορική σημασία. Είναι η πρώτη φορά όπου οι Ευρωπαίοι συνομοθέτες συμπεριλαμβάνουν ρήτρα για την ισότητα των φύλων σε έναν κανονισμό που διέπει ένα ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο. Η διάταξη για την ισότητα των φύλων στον κανονισμό οθείται όσο μας επιτρέπουν οι συνθήκες. Είναι αυτό ένα μεγάλο βήμα, ε, μια νομική καινοτομία που είναι μόνο η αρχή μιας εξέλιξης προς μεγαλύτερη ισότητα των φύλων τα όργανα της Ένωσης. Το Συμβούλιο και το Δικαστήριο και τα κατημέλη δεσμεύονται για την ισότητα των φύλων και δικό μας καθήκον είναι να τους ε, να λογοδοτήσουν μάλλον σε εμά. Κυρία Φεράρα, για ένα λεπτό ευχαριστώ Πρόεδρε. Ας το πούμε ξεκάθαρα. Αυτή η μεταρρύθμιση του δικαστηρίου του Πρωτοβάθμου είναι σκάνδαλο. Στην καλύτερη των περιπτώσεων βρισκόμαστε ενώπιον της προφανούς αδυναμίας του Συμβουλίου Λαϊκού Κόμματος, Σοσιαλιστών και πρασίνων να ξεπεράσουν τη λογική την εθνικιστική που ορίζει ένα κράτος, ένας δικαστής. Όμως ανάγκη είναι να διπλασιαστούν οι δικαστές. Βρισκόμαστε ενώπιον ε, σαφών ε, συμφερόντων για τη μοιρασιά των ε, θέσεων βασικά. Ενώ ζητάμε θυσίες οικονομικές, ε, στην Ιταλία ας πούμε έχουν μείνει μισά ε, τα δικαστήριο. Ενώ εδώ στην Ευρώπη θέλουμε να διπλασιαστεί ο αριθμό των δικαστών. Είμαστε κατά αυτή τη μεταρρύθμιση που προωθεί το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο με ασυνήθιστη βιασύνη. Λυπούμε για του πράσινου και του σοσιαλιστέ, αλλά ούτε καν το φίλο για, τις δίθεν, για την ε, ισότητα των φίλων δεν μπορεί να κρύψει αυτήν την ε, προσπάθεια. Πολύ γρήγορα τα είπατε κυρία Φεράρα. Ο κύριος Λεπρετό. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Αυτή η μεταρρύθμιση είναι σκάνδαλο καταρχήν γιατί είναι άχρηστη. Οι δικαστές που εμείς ε, ακούσαμε στην ε, Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων μας το είπαν, μεταξύ αυτών και ο κύριος Ζάγκερ που είναι και πρόεδρος του Πρωτοβαθμίου. Ε, έχουμε λοιπόν μια μεταρρύθμιση που θα μου κοστίζει 20 εκατομμυριάκια το χρόνο για το τίποτα. Επίσης αυτή η μεταρρύθμιση έχει οδηγήσει σε πολυάριθμες παραβιάσεις της κοινοβουλευτικής διαδικασία του κανονισμού μας για το κανόνα των δύο αναγνώσεων. Η παραβίαση του πιο θεμελιώδους ε, δικαιώματος του βουλευτή που έγινε βιαστικά ε, η ψηφοφορία στις 8 Οκτωβρίου ε, κατά εναντίον μάλλον της άποψης του εισηγητή κυρίου Πίντο. Έπειτα ε, γελίες συνθήκες στη στιγμή που χρειάστηκε με τη βία να μπω στην αίθουσα της Επιτροπής μου που ενώ κάποιοι προσπαθούν να με κρατήσουν εκτός την μέρα της ψηφοφορίας. Παραβίαση δε των συνθήκων της Ένωσης γιατί εκεί προβλέπεται η κατάργηση του δικαστηρίου για ε, του το Δικαστήριο για τη Δημόσια Διοίκηση, οπότε χαιρετίσματα στα δικαιώματα των ε, ευρωυπαλλήλων. Αν θέλετε να τα επαληθεύσετε, έχω και τα συγκεκριμένα άρθρα. Πάντω, όλα δείχνουν τα συμφέροντα των λόμπι και των ιδιωτικών συμφερόντων στην Ένωση. Δεν μα εκπλήσει αυτό, γιατί έχουμε ήδη πολλά παραδείγματα. Ακόμα ένα. Πάντω, 28 θέσει καλοπληρωμένων δικαστών είναι για μοίρασμα. Αυτή είναι το ζουμί. Γι' αυτό το λόγο και είχα θέσει, είχα μάλλον υποβάλει στην Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων μια τροπολογία που απαγόρευε στου ευρωβουλευτέ να γίνουν δικαστέ. Τουλάχιστον έτσι θα θυμίζαμε ένα σοβαρό κανόνα που είναι η διάκριση των εξουσιών, αυτή η τροπολογία ε, περιφθεί. Η πρόεδρος διακόπτη, λυπούμε, τέλειωσε ο χρόνος αγορευσή σας, λυπούμε. Το λόγο έχει η κυρία Κομοντίνη Κάκια. Ευχαριστώ. Χρειαζόμαστε ένα αποτελεσματικό σύστημα δικαιοσύνης Πάντα το χρειαζόμαστε, πρέπει να επενδύσουμε και περισσότερα στο ευρωπαϊκό σύστημα δικαιοσύνης, διότι οι πολίτες χρειάζονται αποτελεσματικό ε, σύστημα δικαιοσύνης. Τι νόημα έχει να δίνουμε σε ευρωπαίους πολίτες το δικαίωμα πρόσβασης στη δικαιοσύνη, στο δικαστήριο και μετά να πρέπει να περιμένουν χρόνια για να αποδοθεί η δικαιοσύνη. Δεν θα πρέπει να απογοητεύονται όσον αφορά τη δικαιοσύνη οι πολίτες θα πρέπει να ε, ε, λύονται διαφορές στο συντομότερο χρονικό διάστημα με δικαστήρια τα οποία θα πρέπει να έχουν καλούς δικαστές και να μπορούν να αποδίδουν δικαιοσύνη. Αυτό περιμένουμε από τα ευρωπαϊκά δικαστήρια. Πράγματι πρέπει να επενδύσουμε περισσότερα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Πάντα αυξάνονται υποθέσεις προς εκδίκαση και δεν βρίσκουν πάντα τις δυνατότητες για να κινηθούν αποδοτικά. Αυτό σημαίνει ότι το δικαστήριο στο οποίο επενδύουμε πρέπει να επαγρυπνεί στο πώς χρησιμοποιεί τους σπόρους του. Θα πρέπει να λογοδοτεί και θα πρέπει να είναι σίγουρο ότι αποδίδεται αποτελεσματικά δικαιοσύνη. Η πρόταση αυξήσεως του αριθμού των δικαστών στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο θα πρέπει να εγκριθεί διότι επενδύει σε αποδοτική δικαιοσύνη για τους πολίτες και δίνει και στο δικαστήριο ε, τη δυνατότητα να αποδίδει δικαιοσύνη. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Δεν θα υπάρξει ε, κόστος για την λειτουργούσα δικαιοσύνη το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο νομολογεί έναντι πολύ μεγάλων ε, επιχειρήσεων παράδειγμα η προστασία δεδομένων από το 10 επί της οποίας υπήρξε η τελευταία πρόσφατη απόφαση. Έχουμε λοιπόν εξαιρετικές αποφάσεις ποιοτικά αναβαθμισμένες. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προσπαθεί εδώ να διασώσει μια απόφαση. Χρειαζόμαστε πράγματι περισσότερους δικαστές. Θα πρέπει όμως να είναι 28 αυτοί οι βουλευτές. Στην ρήτρα αναθεώρησης που απαιτούμε με κάθε σαφήνεια θα πρέπει να επανεξεταστεί το αίτημα αυτό. Και θέλω να υπενθυμίσω το θέμα ισότητα των φύλων. Εδώ μπορεί να διαδραματίσει ρόλο πρωτοπόρου του Ευρωπαϊκού Δικαστήριο. Υπάρχουν τόσες γυναίκες εξαιρετικές ε, δικαστίνες που πρέπει να ληφθεί υπόψη ε, το θέμα αυτό να εκπροσωπούνται ισόρροπα στο ευρωπαϊκό αυτό θεσμικό όργανο. Ευχαριστώ κυρία Τζέιμς για ένα λεπτό. Ακόμα και συγητής βλέπει με κριτικό όμα την πρότασή του. Και έτσι θα πούμε αυτό που έχει υποθεί. Χιούστον έχουμε πρόβλημα. Συνάδελφοι ευρωβουλευτές, έχουμε σοβαρό πρόβλημα. Ακόμα και ο εισηγητής δεν μπορεί να πουλήσει την πρότασή του σε εμά. Ας επιλέξουμε τα σχόλιά του. Βλέπουμε ότι καταδικάζει τα χρήματα, μάλλον περιφρονεί τα χρήματα του φορολογωμένου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει νόμο να αυξήσει τις δαπάνες με αυτόν τον τρόπο. Η νομοθετική αυτή πρωτοβουλία δεν έχει επαρκή διαφάνεια και σε εσωτερικό επίπεδο και σε εξωτερικό. Δεν έγινε ανάλυση κόστους ωφέλους, ούτε ε, εξέταση των συνεπιών. Ζητά απόρριψη της προτάσεως στο τέλος. Τα σχόλια του εισηγητού είναι δικαιολογημένα, ευσταθούν, θα πρέπει να ακολουθηθούν. Απόρριψη είναι η μόνη λύση και το Κοινοβούλιο θα πρέπει να ακολουθήσει τις στάσεις του. Η γιατί στο καλό έχουμε εισηγητές. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μπούντα, για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Επίτροπε αγαπητοί συνάδελφοι. Αναφέρθηκε ότι η καθυστερημένη απόδοση δικαιοσύνης είναι αδικία θέσπιση αδικίας. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να δούμε τον αύξηση του αριθμού δικαστών πρέπει να διασφαλίζεται η ανεξαρτησία των δικαστών, όμως ταυτόχρονα πρέπει να δημιουργούνται μηχανισμοί που θα δημιουργούν την αυθεντική προσπελασιμότητα, την πρόσβαση στην αποτελεσματική δικαιοσύνη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη αυτές τις αρχές ε, και μια ορθή αξιολόγηση των εξελίξεων απαιτείται της προσαρμογής ε, της δομής και της λειτουργίας του δικαστηρίου αυτό θα πρέπει να ανταποκρίνεται στις ε, προκλήσεις που αντιμετωπίζει, που δεν απορρέουν μόνο λόγω του αυξημένου αριθμού κρατών μελών, αλλά και του αυξημένου αριθμού υποθέσεων που εξετάζει το Ευρωδικαστήριο. Πρέπει όλα αυτά να ληφθούν υπόψη και έτσι πιστεύω ότι πολύ γοργότερα πρέπει να λαμβάνονται οι αποφάσεις διότι διαφορετικά υπάρχουν αρνητικές επιπτώσεις με καθυστερήσεις. Η κυρία Γκούτλαντ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύρια Πρόεδρε. Αναμφισβήτητα χρειαζόμαστε περισσότερους δικαστές στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Ο αριθμός των υποθέσεων προς εκδίκαση ε, αυξάνεται και αυτό οδηγεί σε νομική αβεβαιότητα και καθυστερήσεις γιατί δεν εκδικάζονται και κρεμοδικούν. Γιατί επέλεξε αυτή τη θέση το Συμβούλιο, για λόγους πεδαριώδης θα έλεγα. Αλλά για να είμαι ειλικρινή, και τα παιδιά ακόμα θα τα καταφέραν καλύτερα. Ποια είναι η κατάσταση που αντιμετωπίζουμε. Πρέπει να προχωρήσουμε με το όλο χαρτοφυλάκιο, αν θέλουμε τελικά να επομιστούμε τι ευθύνε μα για την ασφάλεια δικαίου. Δεν έχει επιλογή το Κοινοβούλιο. Το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να προχωρήσει. Χρειαζόμαστε όμω να έχουμε και κάποια, κάποιο ποιοτικό επίπεδο στο δικαστήριο. Βλέπετε ότι το ποσοστό των γυναικών στο δικαστήριο είναι μόλι 1%. Νομίζω ότι αυτό είναι προσβολή σε όλε τι ικανέ γυναίκε που κάνουν έξοχη δουλειά στο δικαστήριο. Αρχίζουμε τη διαδικασία Catch the Eye. Έχουμε τέσσερι συναδέλφου να ζητήσουν το λόγο. Ο κύριο Πόσπισιλ θα μιλήσει πρώτο. Ένα λεπτό. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ζήτησα τον λόγο <clears throat> να παρέμβω. Επειδή ήμουν υπουργό δικαιοσύνη στην, δημο... στην ε, Τσεχία και γνωρίζω το τι συμβαίνει με την επιβάρυνση με υποθέσεις των δικαστηρίων, θεωρώ παράλογη αυτή την πρόταση. Διπλασιασμός του αριθμού των δικαστών χωρίς σοβαρή ανάλυση των επιπτώσεων και του αριθμού των υποθέσεων είναι κάτι το ασύλληπτο. Υπολόγισα τι συμβαίνει σε σχέση με το δικαστήριο και είδα ότι υπάρχει αύξηση περιπτώσεων. Όμως αντικειμενικά θα μπορούσε κανείς να αντιμετωπίσει το πρόβλημα με αύξηση, συγκεκριμένη αύξηση του αριθμού των δικαστών. Για παράδειγμα, με αύξηση κατά 10 του αριθμού των δικαστών. Είναι όμως πολιτική απόφαση με βάση κριτήρια που πρέπει να θεσπιστούν γι' αυτό. Όχι όμως ε, απλός διπλασιασμός. Δεν είναι σοβαρό αυτό διότι θα υπάρξουν πολύ μεγάλες επιπτώσεις και χρηματικό κόστος. Έχετε μικρόφωνο κυρία μου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, κυρία Πρόεδρε, είναι μια ένωση δικαίου και το δίκαιο ε, εδράζεται στο δικαστήριο ως ε, υπέρμαχο των δικαιωμάτων των πολιτών και αυτό ε, αποδεικνύεται και από την απόφαση Safe Harbor για τον ασφαλή λιμένα. Μια καθυστέρηση στη δικαιοσύνη είναι αδικία, ναι. Μπορεί να παραμείνει αυτό το σώμα αδιάφορο στα προβλήματα του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου όχι. Τέσσερα χρόνια τα συζητάμε αυτά. Χρειάζεται ένα συμβιβασμό ώστε να είναι πιο αποτελεσματικό το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Υπάρχουν άλλε λύσει. Ναι. Μπορούν να αυξηθούν ε, ε, ο αριθμό των ε, εισαγγελέων, των γενικών δικαστών. Όμω το καλύτερο δεν μπορεί να είναι χειρότερο του καλού ή και του εφικτού και επιπλέον θα πρέπει να υπάρχει διασφάλιση της ισότητας των φύλων για πρώτη φορά με μια διοργανική συμφωνία και δεύτερον μια αναθεωρητική ρήτρα αυτό αξίζει να υπεψηφιστεί. Κύριος Μαριάς παρακαλώ Η αρχή της ευρωπαϊκής συνεργασίας είναι η τήρηση του δικαίου έτσι η ευρωπαϊκή κοινότητα οικοδομήθηκε καταρχάς ως κοινότητα δικαίου μια κοινότητα στην οποία η ερμηνεία και η τήρηση του δικαίου της ανατέθηκε στο δικαστήριό της το οποίο με αποφάσεις κράτησε ζωντανό το ευρωπαϊκό εγχείρημα και άνοιξε νέους δρόμους για την ευρωπαϊκή πορεία. τόσο εγώ όσο και άλλοι καθηγητές διδάσκοντας τους φοιτητές μας στα πανεπιστήμια είχαμε την ευκαιρία να εξάρουμε το ρόλο του δικαστηρίου στην προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών. υποστηρίζω την πρόταση για ενίσχυση του γενικού δικαστηρίου με την αύξηση του αριθμού των δικαστών σε 28 ένας δικαστής δηλαδή ανά κάθε κράτος μέλος προκειμένου να ενισχυθεί έτσι η νομιμοποίηση του δικαστηρίου ενώπιον των λαών της ένωσης να εκπροσωπούνται εκεί ισότιμα όλα τα νομικά συστήματα των κρατών μελών και να καταστεί αποτελεσματική και ταχεία η απονομή της δικαιοσύνης. Ευχαριστώ. Ο Σα ευχαριστώ πρόεδρε. Θα ήθελα κυρίως να ευχαριστήσω επειδή προσπάθησα μια μπλε κάρτα να σηκώσω για να υπάρξει μια παρέμβαση. Δεν το κατάφερα, γι' αυτό θα προσπαθήσω τώρα εκ νέου. Είναι πολύ δύσκολο να κρίνουμε τη δικαιοσύνη σε σχέση με συγκεκριμένες αποφάσεις γνωρίζω ότι υπάρχουν τρόποι να κριθούν ε, οι επιδόσεις της δικαιοσύνης. Όμως για το συμβιβασμό, την εξέβρεση συμβιβασμού όπως, αυτήν, με, όπως αυτόν μεταξύ του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου δεν θα βοηθήσει να επιληθεί η κατάσταση τελικά. Οι δικαστές ε, του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου το απέδειξαν αυτό. Έχω ιδιαίτερε επιφυλάξει όσον αφορά την ψήφιση της πρότασης αυτής. Δεν μπορώ να φανταστώ η μεταρρύθμιση αυτή θα μπορούσε να υποστηριχθεί όπως προτείνεται διότι οι δικαστές του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου ούτε και αυτοί νομίζω ότι ενθουσιοδός διάκυνται. Ολοκληρώθηκε η διαδικασία Κατστιάη και πεθυνόμαστε εκ νέου στην Επίτροπο, την κυρία Κριτσού. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα σχόλιά σας. Ελπίζουμε ότι μπορούμε να στηρίξουμε το συμβασμό μεταξύ Ευρωκοινοβουλίου και Συμβουλίου σαν Ευρωπαϊκή Επιτροπή στον αριθμό των δικαστών στο Γενικό Δικαστήριο και πιστεύω και θεωρώ ότι η δυνατότητα του δικαστηρίου να εκδικάζει τάχιστα τις υποθέσεις και να διευκρινίζονται τα νομικά θέματα γρήγορα είναι κρισίμου σημασίας. Σχετίζεται αυτό και με την πρώτερη συζήτηση που διεξήχθη επί της μεταρρυθμίσεως του εκλογικού συστήματος αφορά την εμπιστοσύνη που υπάρχει μεταξύ πολιτών, των πληθυσμών δηλαδή, και των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Τέλος πάντων, δεν χρειάζεται να το επαναλάβω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλωσορίζει την εξευρεθήσα λύση να προωθηθεί η ισορροπία των φύλων στο δικαστήριο. Αναγνωρίζουμε ότι η ισορροπία των φύλων είναι σημαντική αξία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ εκ νέου. Και νομίζω έτσι θα προλάβουμε να ολοκληρώσουμε και την σύνοδο ε, πριν τα μεσάνυχτα. Ευχαριστώ εκ νέου για τη συζήτηση αυτή. Ο κύριος Μαρίνιο Επίντου για δύο λεπτά. Πρόεδρε, Επίτροπε, εξ ονόματος της αλήθειας της ίδιας δεν είναι αναγκαίοι επιπλέον 28 δικαστές για να επιληθεί οποιοδήποτε πρόβλημα στο Γενικό Δικαστήριο. Αυτοί οι 28 δικαστές ε, είναι μόνο το αποτέλεσμα της ανικανότητας του Συμβουλίου να διορίσει 12 δικαστές που είναι αναγκαίοι σύμφωνα με το ίδιο το δικαστήριο για την επίλυση των προβλημάτων του δικαστηρίου. Από τον Απρίλιο 2014 μέχρι τον Οκτώβριο 2014 από 12 δικαστές περάσαμε στους 28 δικαστές. Αυτό πραγματικά προσβάλλει την ε, ευφυία και την, ε, τις ε, επιδόσεις διανοητικές των Ευρωβουλευτών και των πολιτών της Ευρώπης. Για την ίδια την αλήθεια λέω στο Ευρωκοινοβούλιο ότι οι καθυστερήσεις ε, που παρουσιάζονται δεν οφείλονται σε έλλειψη απουσία δικαστών αλλά σε έλλειψη υπαλλήλων. Κυρία Επίτροπε, είναι διαδικασίες που εδώ και πάνω από ένα χρόνο περιμένουν μεταφράσεις διαδικασίες αναμένουν μετάφραση. Το 2014 εννέα ε, βοηθοί διορίστηκαν. Αυτό έδωσε την δυνατότητα πάνω από 100 δι, ε, υποθέσεις ε, να επιλύονται ανά Εδώ πώς είναι δυνατόν ε, να σηκώσουμε ψηλά τα χέρια εν ώψη του τελεσυγράφου του Συμβουλίου επειδή δεν είναι σε θέση το Συμβούλιο να διορίσει διαφορετικούς δικαστές διαφορετικούς από τον αριθμό των κρατών μελών. Γι' αυτό περνάνε από τους 12 στους 28 ώστε να διορίσουν τους δικαστές τους στα κράτη-μέλη. Αυτό προσβάλλει κατάφορα τα συμφέροντα των Ευρωπαίων πολιτών. Είναι προσβολή στους φορολογούμενους και είναι προσβολή στους στην, ε, στο, στη διανόηση των ίδιων των ε, Ευρωπαίων πολιτών. Δεν είναι αναγκαία αυτά τα κονδύλια και αυτή η αύξηση. Και μάλιστα έχουμε εδώ και έτοιμα τα οποία θα οδηγήσει σε αύξηση κατά 27 εκατομμυρίων ευρώ των δαπανών. Το ε, Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ε, ε, έχει αποτελέσματα μέσα σε τρία χρόνια και όχι σε πέντε. Θα πρέπει να υλοποιηθεί αυτή η μεταρρύθμιση. Κάθε χρόνο έχουμε πάνω από 20 εκατομμύρια ευρώ που θα πληρώνονται ετήσια ενώ θα είχαμε μία εφάπαξ πληρωμή και θα ελύεται το πρόβλημα. Δεν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο σε μία Ευρωπαϊκή Δημοκρατική Ένωση που σέβεται τα συμφέροντα των πολιτών τη. Ευχαριστώ.